Τι θα πούμε στο 1 τρίτο των Ούγγρων που δεν ανήκει στην πλειοψηφία των 2 τρίτων. Τι θα του πούμε, ότι δεν πρόκειται να έχουν ποτέ ξανά ευκαιρία μετά τι επόμενε εκλογέ να ε, τροποποιήσουν το σύνταγμα αυτό και τι μεταρρυθμίσει. Ευχαριστώ. Για την ομάδα της αριστεράς, κύριος Ταβάρες, για δύο λεπτά.